Good morning, ladies and gentlemen. May Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Okay, I open... Λοιπόν, κηρύσω την άναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και αρχίζουμε με την έγκριση της ημερησίας διάταξης, παρακαλώ. Εγκρίνεται το σχέδιο ημερησίας διάταξης ή έχετε κάποια πρόταση ή αλλαγή. Όχι, ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, δεν έχω ανακοινώσει σήμερα. Ελπίζω μετά την συνεδρίαση των συντονιστών θα έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις και κάτι θα έχουμε να σας παρουσιάσουμε ως ανακοινώσεις ε, της Πρόεδρου, αλλά αυτό θα είναι για μετά. Και έτσι φτάνουμε τις κατ' ουσίαν συζητήσεις μας και ξεκινάμε με μια πολύ σημαντική έκθεση που είναι η πολιτική συνοχή και ο θεματικός στόχος για την προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και την εξάλληψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων. Η εισηγητής μας είναι ο κύριος Νοβάκοφ. Έχουμε και τους σκιώδες εισηγητές εδώ, έχουμε και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Νοβάκοφ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης και σας το λέω και τώρα θα το πω και στο τέλος ότι προτείνουμε την 26η Φεβρουαρίου ως προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι το τέλος της ημέρας, έτσι. Λοιπόν, κύριε Νοβάκοφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα στους συναδέρφους. Δεν είμαι γιατρός, ποτέ δεν πήγα να παρακολουθήσω μαθήματα ιατρικής, ποτέ δεν θα ξέρα πώς να αντιμετωπίσω έναν ασθενή. Ξέρω όμως τι κάνουν οι γιατροί για να βοηθήσουν. Και το πρώτο που κάνουν είναι ότι κάνουν τη διάγνωση. Οπότε είμαι περήφανος που έχω την ευκαιρία να εκτιμήσω το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η πολιτική συνοχή για να βελτιώσει τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι είναι εντυπωσιακή εικόνα. Γιατί παρόλο που δεν καταφέραμε να στείλουμε ένα αυτοκίνητο στο διάστημα, χάρη στην πολιτική συνοχής, ε, Παρ' όλα αυτά όμως εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ οι πολιτική συνοχή και όσοι πιστεύουν σε αυτή, καταφέραμε να βελτιώσουμε τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ. Και οι βελτιώσεις αυτές είναι τόσο μεγάλες που κανένας δεν ε, είχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα δεν θα ήθελα εδώ να σας γεμίσω νούμερα που έχω χρησιμοποιήσει για να καταλάβω γιατί είναι τόσο σημαντική η πολιτική αυτή και γιατί οι επενδύσεις στις μεταφορές επηρεάζουν τόσο πολύ τη η καθημερινότητα των ανθρώπων. Αν βγείτε από αυτή την αίθουσα και πάτε στον αυτοκινητόδρομο προ το Βατερλό, θα δείτε αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία. Ναι, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι στα οχήματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο γυρνάει από τη δουλειά του πίσω στην οικογένειά του με ασφάλεια. Ε, είναι κανείς σε θέση αυτό να το αξιολογήσει, να το εκτιμήσει σημαίνει επίσης ότι έχουμε πολύ λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, επειδή είναι καλύτερη η δρόμη μας. Αυτό το εκτιμάμε. Πόσες ζωές σώζονται επειδή είναι καλύτερη η δρόμη μας. Δεν αξιολογείται όμως αυτό επαρκώς. Οπότε θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε ποσοτικά αυτές τις βελτιώσεις. Όμως, το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να στροφακαμιλίζουμε και να παραβλέπουμε άλλες πρωτοβουλίες ανά το κόσμο όταν πρόκειται για τις μεταφορές. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Και ξέρω ότι βρισκόμαστε στην κρίσιμη καμπή, όπου πρέπει να αποφασίσουμε πόσο θα παιδίσουμε σε άλλες πολιτικές και στις μεταφορές και ξέρω ότι θα κοστούν πολλές φωνές που θα υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη πολιτική. Όμως οι μεταφορές αναφίβολα, είναι από τις πολιτικές που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο μέλλον, όποιο και αν είναι το τίμημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Μια από τις πρώτες χώρες που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποχωρεί. Και αυτό είναι ένα σοκ για όλους μας. Χάνουμε έσοδα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε και κυρίως στις χώρες εκείνες που μπήκαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που εξαρτώνται πραγματικά από τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Οι επενδύσεις μακριά από τις Βρυξέλλες δεν βοηθούν μόνο τον τοπικό πληθυσμό εκεί. Μην ξεγελιόμαστε οι γέφυρες που συνδέουν τη Βουλγαρία με τη Ρουμανία στο Δούναβι δεν βοηθούν μόνο τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί είναι πάρα πολλά φορτηγά από την Πολωνία, ε, το Βέλιο, τη Γερμανία, που περνάνε από τέτοιες γέφυρες. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν είμαι γιατρός και ίσως πολλοί από εσά αναρωτιέστε καλά γιατί ξεκίνησε έτσι. Όμως τα δίκτυα μεταφορών παρουσιάζουν την ίδια εικόνα όπως είναι το κυκλοφοριακό σύστημα σε έναν ανθρώπινο οργανισμό. Για να έχουμε λοιπόν έναν ευρωπαϊκό οργανισμό υγιή, χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό κυκλοφοριακό σύστημα. Άρα η συμφόρεση είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Και ναι, το λέω αυτό γιατί όντως κάθε περιφέρεια πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο μέσο όρο της ευημερία. Ε, αλλά συγχρόνως πρέπει να επενδύουμε και αρκετά στα οδικά δίκτυα. Τι έχουμε καταφέρει λοιπόν μέχρι τώρα. Ακριβώς εξαιτίας των επενδύσεων, κυρίως διασυνοριακά, των επενδύσεων στα οδικά δίκτυα, πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες έχουν μειώσει το χρόνο που χρειάζονται για να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο. Για να μην πω και πόσες ζωές έχουν σωθεί εξαιτία της βελτίωσης των οδικών αυτών δικτύων. Οπότε αυτό που κάνει η έκθεσή μου, τώρα μάλιστα, πριν αρχίσει η συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, πρέπει να κάνουμε τη διάγνωση πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Προς το παρόν είναι η πολιτική που κυριαρχεί. Εγώ θα ήθελα περισσότερο οικονομία όταν μιλάμε για μεταφορές. <clears throat> Και ξέρω ότι είναι περίεργο να το λέμε αυτό σε ένα πολιτικό σώμα, όμως, όταν μιλάμε για σιδηροδρόμους, για αυτοκινητοδρόμους, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να εντοπίσουμε που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Και όταν είμαστε στα διευρωπαϊκά δίκτυα, να μην ε, μπερδευόμαστε με διαφορετικές πολιτικές εντάσεις, ιδεολογίες, πολιτικές κτλ. Δεν είναι αυτά που πρέπει να κυριαρχούν στη συζήτηση. Γιατί όλοι μας εδώ καταλαβαίνουμε γιατί είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να πάει από το Άμστερνταμ στην Βάρνα από αυτοκινητόδρομο. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό για τις επιχειρήσεις, πόσο σημαντικό είναι για τους τουρίστες, για τις υπηρεσίες, για τους ανθρώπους. Στην Αφρική υπάρχουν πάνω από 50 χώρες. Και αν ρωτήσετε τους πολίτες των χωρών αυτών ποιοι είστε, τι θα πούνε, θα πούνε είμαι Αφρικανό. αυτό θα είναι το πρώτο που θα πούνε. Και μετά θα πούνε από ποια χώρα προέρχονται. Και εγώ έχω ένα όνειρο, όταν πηγαίνουμε στι διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ρωτάμε κάποιον ποιον είναι, να λέει πρώτα ότι είναι Ευρωπαίο και μετά ότι είναι Βούλγαρο, Τσέχο, ε, Πολωνό κτλ. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν έχουμε καλούς δρόμους, καλές μεταφορές. Και όσο και αν ο κόσμος μας γίνει ψηφιακός στο μέλλον, παρόλα αυτά πάντα θα χρειαζόμαστε καλύτερους αυτοκινητοδρόμους, ε, μεγαλύτερα λιμάνια, αεροδρόμια και πιο γρήγορα τρένα. Ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, οπότε δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προτεραιότητα αυτή. Και πιστεύω ότι αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα είναι υπέροχα. Και κανείς στην ανθρώπινη ιστορία δεν έχει καταφέρει εν καιρό ειρήνης, να πετύχει τόση αλληλεγγύη μεταξύ ανεξάρτητων χωρών σε τέτοιο επίπεδο και είναι προφανές το αποτέλεσμα. Αναφερθήκαν οι προθεσμίες. Μπορούμε να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης για τη συνεισφορά της συνοχής και των διαφορετικών ταμείων στα δίκτυα μεταφορών. Οπότε πιστεύω ότι όλοι θα στηρίξουμε αυτή την θέση για να διασφαλίσουμε ακριβώς ότι η Επιτροπή μας θα εισακουστεί σε μερικούς μήνες όταν θα αρχίσει η συζήτηση για το πόσα χρειαζόμαστε για τις μεταφορές μετά το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Νοβάκοφ. Και τώρα ο λόγος στους και ηγητές. Μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζωτόφσκι που εκπροσωπεί σήμερα εδώ την Επιτροπή Μεταφορών. Η Επιτροπή Μεταφορών αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση με βάση το άρθρο 53 συν ε, για την έκθεση αυτή. Από ό,τι σήμερα ο κύριος Ζωτόφσκι θα μας παρουσιάσει την θέση της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Αφού όμως ακούσουμε τους σκιώδης ηγητές πρώτα, οι σκιώδης ηγητές όμως ο κύριος Πίτσουλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και αρθρωτικών ε, ταμείων συνέβαλαν στη βελτίωση και των περιφερειών και της κατάστασης των χωρών μελών και περιόρισαν τον αριθμό της. Για παράδειγμα, σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, από τα 7.500 ε, μέτρα νέα σιδηροδρομικό γραμμό να κατασκευαστούν. Και το πρώτο ήταν για την ανανέωση. Θα πρέπει επίση να δώσουμε έμφαση στη διασυνοριακή διασύνδεση. Για παράδειγμα, τα λιμάνια, προδρομικές γραμμέ, τα ίδια μέτρα ε, θα πρέπει να τα υιοθετούμε και για τα λιμάνια. Και μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί, διάδρομοι έμειναν κατά 80% να αυξηθούν οι εμπορικές μεταφορές και ε, κατά 60% οι μεταφορές επιβατών, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε στο κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό και θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και ε, κύριε, εκ μέρους του κυρίου Πορέμπα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, συντάκτη της, της έκθεσης, τον κύριο Νοβάκοφ Επίσης, περισσότερο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και ήδη είχαμε πολλά επιτεύγματα στον κλάδο αυτό. Ε, Διαφορετικό ο ρυθμό ανάπτυξη των υποδομών μεταξύ Δυτικής και Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα παρόμοιο ε, ρυθμό ανάπτυξη και ποιότητα υποδομών. Και σίγουρα είχαμε από τη Θράκη μέσω του Μαυροβονίου και ε, στον Μπουργά δημιουργήθηκε ένα ο σχετικός αυτοκινητόδρομος ή ε, υποδομών μεταφορών. Χρειαζόμαστε καλό οδικό δίκτυο, εξυγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί από όλα αυτά θα εξαρτηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον Είναι μια πιο σφαιρική ανάλυση του οικονομικού μοντέλου, της παγκοσμιοποίησης, της ανταγωνιστικότητας ενιαίας αγοράς, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για τις υποδομές που θα πρέπει να έχουν καλύτερες ικανότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερες και πιο ποιοτικέ υποδομές και φυσικά αηφόρες υποδομές. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες αλλαγές παρόλα αυτά που να μειώνουν την ανάγκη των υποδομών, κάνοντας ένα παραλληλισμό ε, με αυτό που λέμε ότι η πιο βιώσιμη αηφόρος ενέργεια είναι αυτή που δεν ε, καταναλώνεται. Θέλουμε λοιπόν ένα πιο ισορροπημένο και αποκεντρωμένο οικονομικό μοντέλο που θα περιορίζει τη τεράστια μεταφορά ε, εμπορευμάτων και ε, εργαζομένων και θα μειώνει τις ανισότητες μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρων ή τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της αστιφιλίας και της απερίμωσης άλλων ζωνών αναφέρθηκαν στην έκθεση και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του σχεδίου Juncker ε, και των ε, συμπράξεων ε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δίνουν εγγυήσει δημόσιου χαρακτήρα στι ιδιωτικέ επενδύσει. Θα πρέπει να κινητοποιούμε και ιδιωτικά κονδύλια, όχι μόνο δημόσια κονδύλια, αλλά αυτό να μην γίνεται ει βάρο των κονδυλίων που καλό θα είναι να εξυπηρετούν στους πολίτες. Στην Ισπανία είχαμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια που αφιερώθηκαν για τη διάσωση των αυτοκινητοδρόμων και αυτό έγινε που είχαν γίνει με ιδιωτικά κονδύλια, ενώ αυτή τη διάσωση θα την πληρώσει τώρα ο Ισπανός φορολογούμενος, ο Ισπανός πολίτης. Επίσης, ε, ε, δεν θα πρέπει κάποιοι ιδιώτες ε, να διακινδυνεύουν τα χρήματά τους με δημόσιες εγγύησεις γιατί δεν θα πρέπει με δημόσια κονδύλια να καλύπτουμε τις ζημίες ή τον κίνδυνο των ιδιωτών επενδυτών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις βιώσιμες μεταφορές με υψηλότερη κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, ε, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων με άμεση συμμετοχή και δυνατότητα συναπόφασης των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Έτσι, τα έργα υποδομής θα είναι πραγματικά ε, το αποτέλεσμα πραγματικού δημοσίου διαλόγου, μελέτης ε, και κοινωνικών αλλά και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολύ εύστοχα λέει η έκθεση ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες τονίζοντας την ανάγκη της ε, διαπεριφερειακής συνεργασίας και της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ε, μεθόριων περιοχών. Επίσης, ε, με τις επιχορηγήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δημόσιες μεταφορές επιβατών και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους σιδηροδρόμους και για τη μεταφορά εμπειρευμάτων και για τη μεταφορά επιβατών, γιατί οι σιδηρόδρομοι είναι το πιο βιώσιμο μέσο μεταφοράς και το πιο φιλοπεριβαλλοντικό, το λιγότερο ρηπογόνο. Επίσης, έχουμε εγκαταλειμμένες ε, συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το μεγάλο δυναμικό που έχουν για τη διαφύλαξη του εδαφικού και, περιφε... κοινωνικού ιστού και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απερίμωσης περιοχών. Επίσης, ε, θέλουμε οι μεταφορές μας να συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμφωνίες της COP21 των Παρισίων. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, στη βιωσιμότητα των μέσων μεταφοράς και στην ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τους αυτοκινητοδρόμους, ώστε να τους καταστήσουμε πιο ασφαλείς και να περιορίσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Και επίση να μην ξεχνούμε την ποιότητα τη απασχόληση και τι κατάλληλε εργασιακέ συνθήκε των εργαζομένων που συμμετέχουν σε έργα υποδομή μεταφορών, λαμβάνοντα υπόψη και τηρώντα ε, τι ε, επόμενε μα ε, συζητήσει και συναντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ροπ, εκ μέρου του Σκιώδου, εισηγητή στόχος για όλα τα κράτη-μέλη και να πιστούν οι πολίτες μας ότι χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους καθαρές πηγές ενέργειας στις μεταφορές τους συμβάλλουν ε, και νομίζω ότι ε, μέσω της συζήτησης που θα έχουμε θα καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λοτόφσκι για να μας παρουσιάσει τη θέση οδηγούς φορτηγών και τις γερμανικές επιχειρήσεις που στέλνουν τα φορτηγά τους από τις υποδομές αυτές. Συνεπώς, με τις επενδύσεις πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα ανά την Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές υποδομές είναι ο καλύτερος τρόπος να επενδύσουμε. Έχουμε ε, την καλύτερη απόδοση, γιατί κάτι το οποίο φαίνεται να είναι τοπικό, τελικά όμως μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις διευρωπαϊκά. Η επένδυση που έγινε στις ε, συμφορήσεις είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομίες περιφερειών πολύ λιγότερο ευνοημένες που μπορούσαν ναι, να έχουν πρόσβαση στη μάχη κτλ. Ας μην πω σε λεπτομέρειες. Συνεπώς, οι επενδύσεις για να αποφεύγονται συμφορήσεις στις υποδομές μεταφορών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτές οι συμφορήσεις δημιουργούν και ανισότητες τοπικά και που δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι συμφορήσεις. Και εκεί που έχουμε πραγματικές συμφορήσεις πρέπει να κοιτάξουμε πολύ καλά τα στοιχεία. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολες περιπτώσεις. Και όταν επενδύουμε μπορεί μεν να αποδίδουν, αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι συμφορήσεις, δεν βλέπουμε στην πραγματικότητα πώς επηρεάζουν ε, τα... την κατάσταση γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να περάσουμε έτσι κι αλλιώς από τις οροπορικές δρομικές μεταφορές. Το έχουμε πει αυτό που είναι περισσότερο βιώσιμες και πολύ χαίρομαι για το παράδειγμα που έδωσε ο συνάδελφος εδώ πίσω μου για το πώς μπορούμε να περάσουμε ε, από τους σιδηροδρόμους στις πράσινες μεταφορές. Θέλουμε πιο βιώσιμα οχήματα, περισσότερο ηλεκτρικά οχήματα, πιο πράσινα. Οι επενδύσεις στις οδικές υποδομές στο μέλλον θα περάσουν και από επενδύσεις που κάνουν πιο πράσινο το δρόμο, πιο πράσινες τις οδικές μεταφορές, πιο οικολογικές. Αυτό είναι οικολογικά οχήματα. Χαίρομαι λοιπόν για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι μπορεί πράγματι να βελτιώσει τη σκέψη μας. Εγώ θα υποβάλω μια-δυο επικοδομητικές τροπολογίες, αλλά κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τον εισηγητή και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστούμε κύριο Φανίστερο, είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρουσίαση που είχαμε σήμερα το πρωί και για τόσα ακούσαμε μέχρι τώρα από πλευρά του ΕΛΚ που ζήτησε την έκθεση αυτή. Είναι μια εφαρμοστική έκθεση, έτσι, το πώ δηλαδή εφαρμόζονται τα πράγματα, δεν είναι καθαρά μια έκθεση πολιτικής. Εξετάζουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι 81 δισεκατομμύρια δαπανώνται από τα ταμεία μας, συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και πρέπει να το πούμε ότι η προτεραιότητα παρέμεινε αυτή την περίοδο. Πολλά αλλάξαν, οι θεματικές συγκεντρώσεις, σε γνώση, διάδοση γνώσης, διάδοση της γνώσης λοιπόν, αλλά παρέμεινε αυτή η προτεραιότητα και είναι σημαντικό να το πούμε ότι η πολιτική μεταφορών εξακολουθεί να βασίζεται στη συνοχή. Την προηγούμενη περίοδο αποφάσισε η Επιτροπή μας Περιφερικής Ανάπτυξης για τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία πήγαν τελικά στην ε, ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Και οι χώρες μπόρεσαν να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά με δικές τους προτάσεις μέχρι το 2018, έτσι. Και τώρα θα έπρεπε να αποκτήσει πιο κεντρικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ είναι που είδαμε πολύ θετικές επιδράσεις, γιατί χώρες τράφηκαν πιο πολύ διασυνοριακά πολύ περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη περίοδο. Οπότε θα μπορούσαμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες προκειμένου ε, το σύστημα αυτό στην επόμενη περίοδο, πέρα από τη συνοχή, όπως είπατε κι εσείς, να μπορεί να αφοσιωθεί προκειμένου να διατηρηθεί αυτός ο μηχανισμός. Να είμαστε πολύ κοντά στην ε, Επιτροπή Μεταφορών και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε από το παρελθόν. Αλλά όχι να πούμε όχι βάλτε τα χρήματα στην ε, διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Όχι. Θα πρέπει να συνδέσουμε τα δύο μέσα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρξει αυτή η συνέργεια μεταξύ τους. Είναι ακριβώ αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, Αντρέη Νόβακοφ. Αν υπάρχει σύνδεση, μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο την οικονομία. Αν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, δεν μπορείτε να αποτελέσετε ένα πόλο ανάπτυξη. Οπότε στο πρώτο στάδιο, μετά την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταφορές ήταν νούμερο ένα και παραμένει. Αλλά ίσως χρειάζεται περισσότερη διαφοροποίηση στο μέλλον. οδικές μεταφορές και συνδρομικές μεταφορές. Ας το σκεφτούμε. Ε, θα διατηρήσουμε το σύστημα αυτό της διευκόλυνσης ιδέοντας στην Ευρώπη. Το θέλουμε. Ε, εγώ θα έλεγα ναι. Και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην έκθεση, τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει για να περάσει στη συνέχεια και στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τον κύριο Λάινερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο ευχαριστώ πολύ που έχουν υποστηριχθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο πιο θετικά σχετικά με, το, με τα ποσοστά και τους ρυθμούς επιλογής προγραμμάτων και έργων ε, που αφορούν στις ε, μεταφορικές επιδομές. Το 2017 στο τέλος ο ρυθμός επιλογής έργων ε, ήταν πάνω από 61% για επενδύσεις στα TNT το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 64% και για τις επενδύσεις ε, στους αεροδρόμους του βασικού δικτύου TNT το ποσοστό ήταν 66% μάλιστα. Ε, νομίζω ότι στα τέσσερα χρόνια εφαρμογής ε, του προγράμματος ε, τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά ενθαρρυντικά και θετικά. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για τις διευκρινήσεις αυτές. Αυτά λοιπόν ήταν τα σχόλια επί του σχεδίου έκθεσης. Κύριε Νοβάκοφ, έχετε το λόγο για να κάνετε τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις και να απαντήσετε αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα όλους τους συναδέλφου και νομίζω ότι αυτό είναι και η ομορφιά αυτής τη Επιτροπής μας. Ακριβώς δηλαδή η δυνατότητα που έχουμε να εκφράζουμε και να ακούμε διαφορετικές απόψεις από το τη Ένωση έως και την, το άλλο άκρο του φάσματος ε, ε, που αναφέρει ότι χρειαζόμαστε απολύτω και του ιδιώτε επενδυτέ προκειμένου να επιτύχουμε του στόχου μα. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η αλήθεια μάλλον θα βρίσκεται κάπου στη μέση. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Κύριε Χάουαρντ, θα ήθελα να ξεκινήσω με τα δικά σας σχόλια. Εκτιμώ πολύ αυτά που είπατε και νομίζω ότι ενίσχυσε και την άποψή μου ε, όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζω εγώ την πολιτική. Αν χάσει κανείς το προκειμένου να ε, ολοκληρώσουμε το δίκτυο TNT. Με προϋπολογισμό 22 δισεκατομμυρίων στο ΣΕΦ, νομίζω ότι πόρο απέχουμε από το να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή μας να καταφέρει να ασκήσει πίεση και είδους προγραμμάτων όπως το Connecting Europe Facilities για τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να αρχίσουμε να εξηγούμε και χωρίς να ε, κάνουμε την κλασική συζήτηση για συνεισφέροντες και αποδέκτες ε, κονδυλίων. Δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε σε αυτή τη συζήτηση συνεχίζω ότι δεν είναι πάντα ένα συν ένα μας κάνουν δύο, κάποιες φορές μας κάνουν και τρία και τέσσερα. Άρα, ένα μεγαλύτερο προπολογισμό για το ΣΕΦ θα είναι μια καλή αφιτηρία. Το να εξασφαλίσουμε λοιπόν επαρκή χρηματοδότηση για την ε, συνοχή είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία πρέπει να χαράξουμε και να υπερασπιστούμε όσο το δράσπιση της ε, πολιτικής συνοχής. Προσβλέπω λοιπόν με μεγάλη χαρά στη συνεργασία με όλους σας και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε, ε, μια, σε ένα καλό κείμενο να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι στην Ευρώπη που δεν θα κατα... αν ένας ελικιωμένος δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακά του ακόμα και αν δεν είναι παππούς μας ή γιαγιά μας. Αυτά είναι τα θέματα που μας, πρέπει να μας απασχολήσουν. Είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη όλα αυτά τα θέματα. Είμαι ανοιχτό στη συζήτηση, στις τροπολογίες που θα καταθέτεις και σας ευχαριστώ Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ψηφοφορία επί της έκθεσης θα γίνει τον Μάρτιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ξέρετε ότι η 7η αυτή η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου που μας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την μας Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας προκειμένου να παρουσιάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη της μεταρρύθμισης αυτής. Ορίσαμε το τμήμα πολιτικής Β και την 1η Φεβρουαρίου είχαμε μια εκτακτή συνεδρίαση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μετά δηλαδή το 2000. Είναι 5 ώρα το απόγευμα, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Θα σας το υπενθυμίσω και στο τέλος της συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα συζητήθηκε όντως ξανά. Είναι μια σημαντική υπόθεση και είναι αλήθεια ότι αυτό που του δίνει ιδιαίτερη διάσταση είναι ότι η έκθεση αυτή μας έρχεται σε μια στιγμή κλειδί. Μετά δηλαδή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μελλοντικό προπολογισμό και για τα διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2020. Η Επιτροπή μας λοιπόν έχει ήδη την ευκαιρία να τοποθετηθεί για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Κυρίως με την έκθεση του συναδέλφου πάλι και εννοείται ότι συμφωνώ με την συνέχεια των εργασιών του. Στο μεταξύ βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν προχωρήσει και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και διάφορα στοιχεία τα οποία είναι νέα κυρίως την 7η έκθεση συνοχής που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να συντάξω την έκθεσή μου προσπάθησα να συμβιβάσω διάφορους στόχους. Να πάρουμε μαθήματα από την έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα και θα επανέλθω σε αυτό. Είναι πολύ πλούσιο το έγγραφο αυτό, πυκνό, πλήρες και αντικατοπτρίζει το έργο όσων συμμετείχαν. Όμως δεν ήθελα να έχω μία έκθεση που να είναι απλά ε, περιγραφική, που παρουσιάζει απλώς στοιχεία. Η προτεραιότητά μου είναι να πάρουμε τα μαθήματα από αυτή την 7 έκθεση συνοχής για να καταλήξουμε σε προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και ο τρίτος στόχος μου ήταν να περάσω και ένα πολιτικό μήνυμα για να υπενθυμίσω διάφορες αρχές που πιστεύω ότι είναι βασικές. Τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος για να στηρίξουμε την πολιτική συνοχής, για να στηρίξουμε μια πολιτική συνοχής δηλαδή που να είναι φιλόδοξη. Και πρέπει όλοι μαζί να αντιταθούμε όσο μπορούμε περισσότερο με πυγμή σε κάθε σενάριο το οποίο θα οδηγούσε να αποκλειστούν κάποιες περιφέρειες ή κάποιες χώρες από την μελλοντική πολιτική συνοχής. Κατά τη γνώμη μου ένα είναι το σενάριο που θα πρέπει να υπάρχει και αυτό είναι μια πολιτική συνοχής που να καλύπτει το σύνολο των περιφερειών των ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε, για να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από τα μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε. Η Επιτροπή συχνά τονίζει την προστιθέμενη αξία. Κάθε σελίδα της έκθεσής της υπογραμμίζει αυτήν την προστιθέμενη αξία, είναι αλήθεια. Και προσπάθησα και εγώ να προσεγγίσω το θέμα υπογραμμίζοντας ότι η έννοια αυτή της προστιθέμενης αξίας εμφανίζεται από την πολιτική συνοχή η οποία προσπαθεί να φέρει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της. Μια άλλη βασική αρχή, η οποία υπογραμμίζεται στην έκθεση της Επιτροπής, είναι ότι ο αντίκτυπος αυτών που όλοι γνωρίζουμε, από, όπου, από ποια χώρα και αν δηλαδή της παγκοσμιοποίησης, της επιτάχυνσης της παγκοσμιοποίησης, της φτώχειας, της κλιματικής αλλαγής, όλες αυτές ε, Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό και στηρίζω μια πολιτική συνοχή η οποία θα συνεχίσει να καλύπτει το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών, χάρη βέβαια σε έναν προπολογισμό που θα μας γίνει γνωστός, αλλά που θα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους των προκλήσεων. Και έπειτα, αν πρέπει να καλυφθούν όλες οι περιφέρειες, εδώ η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ε, σε ποιο σημείο ε, διαφέρουν οι ανάγκες των ε, περιοχών μέσα στην Ένωση. Και σε αυτό το πλαίσιο η εδαφική διάσταση της πολιτικής ε, συνοχής πρέπει, πιστεύω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου, να ενισχυθεί περισσότερο. Και αυτό για να εξασφαλιστεί μία προσέγγιση που να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη. Και αυτό για όλες τις ε, περιφέρειες, είτε πρόκειται για παραμεθόρειες, είτε πρόκειται για άκρος κτλ. Πρέπει να μειωθούν οι διαφορές που υπάρχουν. Η έκθεση δείχνει επίση ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, ότι υπάρχουν αντιφάσεις μερικές φορές, ότι υπάρχουν ε, διαφορές οι οποίες μάλιστα οξύνονται ή μετατοπίζονται. Η έκθεση, για παράδειγμα, υπογραμμίζει ότι υπάρχουν θύλακες ένδυας, ότι υπάρχουν ε, περισσότερες διαφορές ε, διαπεριφερειακά ακόμα και μέσα σε πλούσιες περιφέρειες. Επίσης δείχνει ότι το επίπεδο ανεργίας παραμένει υψηλό σε σχέση με πριν από την κρίση και ένα άλλο μάθημα που παίρνουμε από αυτή την έκθεση και το έχουμε ήδη συζητήσει εδώ είναι η περίπτωση περιφερειών που τις ονομάζουμε εγκλωβισμένες στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματος. Το έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, είχαμε εξηγήσει για αυτό το φαινόμενο των περιφερειών που είναι εγκλωβισμένες στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματος. Κατά τη γνώμη μου, πολλά διακυβεύονται για την μελλοντική πολιτική συνοχή. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε απαντήσει, να δώσουμε λύσει για τι περιφέρειες αυτές. Η πολιτική συνοχή δεν πρέπει μόνο να μειώσει τις διαφορές, πρέπει επίσης να προβλέψει και να προλάβει την απομάκρυνση κάποιων ε, περιφερειών που είναι έθραυστες. Αυτό όσον αφορά τα μαθήματα, τα κύρια μαθήματα δηλαδή που παίρνουμε από αυτήν την έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο. Αλλά τώρα βάσει των μαθημάτων αυτών της 7ης έκθεσης προσπαθώ να κάνω και προτάσεις προκειμένου οι επισημάνσεις αυτές να αντικατοπιστούν στην νέα πολιτική συνοχής. Και γι' αυτό επέλεξα κάποιες προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις παραβάσεις. Εγώ προτείνω μια θεματική συγκέντρωση, ισχυρή θεματική συγκέντρωση, η οποία να βασίζεται στους μεγάλους στόχους, όπως συμβαίνει με τους μεγάλους πολιτικούς στόχους ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Απασχόληση, καινοτομία, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και κλιματικές αλλαγές. Αντίθετα, όχι σε βάρος της εδαφικής προσέγγισης, που έτσι κι είναι πολυθεματική από μόνη της. Πιο περίπλοκη και στην οποία πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Οπότε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακέ περιφερειακές διαφορές. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό όπως σας είπα. Τώρα όσον αφορά τους δείκτες. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτούς. Το βασικό είναι ότι οι νέοι δείκτες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μέρος της πολιτικής συνοχής. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το Ταμείο αυτό έχει μια εδαφική διάσταση. Κάναμε στρατηγική σημασία λάθος. Και τέλος, για ένα θέμα γενικά ευαίσθητο. Πιστεύω ότι οι προτεραιότητές μας και τους στόχους μας. Πιστεύω επίσης ότι είναι αναγκαίο πρέπει να ασχοληθούμε με ζητήματα όπως είναι η σύνδεση της συνοχής με την κοινωνική και φορολογική σύγκληση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να κινδυνεύσουν ακόμα περισσότερο κάποιες ε, έθραυστες εδαφικές οντό. Βάλουμε μια νέα αρισιμότητα, νέες προϋποθέσεις που είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, ούτε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να Τέλος, κάτι άλλο το οποίο όλους μας απασχολεί πολύ και στο οποίο έχω δώσει κι εγώ μια πέρια και όπου συμμετέχουν όσοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες ήδη παγικότητα και η διαφοροποίηση. Αυτά λοιπόν με λίγα λόγια, ποιες είναι οι βασικές γραμμές της έκθεσής μου που σας προτείνω αδέρφου και σκιώδες εισηγητές. Για να τηρηθεί όμω το χρονοδιάγραμμα αυτό, παρακαλώ τους συναδέρφους να υποβάλουν τι τροπολογίε του στα αγγλικά. Αν... Thank you very much. You are right. ευχαριστούμε κύριε Ζούλο. Όντω, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να εκπονήσουμε την έκθεση και να τη δημοσιεύσουμε πριν το σχέδιο το του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, και λυπούμε που θα μακρηγορήσω λίγο, αλλά όντως η έκθεση είναι και πολύ σέλιδη αλλά και πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας πάντως ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αξιόλογη έκθεσή του ε, σε μεγάλο βαθμό άλλωστε συμφωνούμε μαζί του και θα ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή του για επίσπευση των συζητήσεων και των προσπαθειών ώστε να καταφέρουμε να υποβάλουμε την έκθεσή μας στην Ολομέλεια πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει τις προτάσεις της για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια γενική παρατήρηση, ένα γενικό σχόλιο. Ε, κάποια τμήματα της έκθεσης ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα στην, ε, στις αιτιολογικές σκέψεις, που πιστεύω ότι καλό θα ήταν να περάσουν από το αιτιολογικό στο διατακτικό, γιατί στο τελικό κείμενο δεν προσέχει κανείς τις αιτιολογικές σκέψεις, ενώ μερικές είναι πολύ εύστοχες και καλό θα ήταν να περάσουν στο διατακτικό. Οπότε είτε ο ίδιο ο εισηγητή, ίσω μέσω, των τροπολογιών θα μπορούσαμε κάποια εύστοχα στοιχεία των αιτιολογικών σκέψεων να τα μεταφέρουμε στο κυρίως τμήμα, στο διατακτικό της έκθεσης. Ακολουθώ τώρα τον Ιρμό και τη σειρά των σημείων του εισηγητού και να πω ότι φυσικά συμφωνούμε με τη θέση ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και επίσης το γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκυται ακριβώς ε, στην επικουρικότητα και στην ε, ανάμειξη και των περιφερειών στην εκπόνησή της και έτσι έχει την ικανότητα και εκεί έγκυται η προστιθέμενη αξία στο να φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Αυτό ίσως ε, δεν αναγνωρίζεται δεόντως την παρούσα συζήτηση για την πολιτική συνοχή που έχει την τάση να επικεντρώνεται στα αρνητικά σημεία και σε κάποιες καθυστερήσεις που σημειώνονται. Γι' αυτό και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις της πολιτικής συνοχής οφείλονται σε μια ε, εσφαλμένη αντιπαράθεση. Γιατί θεωρούμε ότι τα, ταμεία του τα κονδύλια του Ταμείου σχεδίου, ε, Juncker, του Σχεδίου Juncker δίνονται όταν ε, προβλέπονται τα κονδύλια, αλλά στη συνοχή θεωρούνται τα αποτελέσματα ορατά μόνο όταν ολοκληρώνονται ε, τα προγράμματα. Οπότε σε αυτή την ασφαλμένη αντιπαράθεση οφείλεται η εντύπωση ότι η πολιτική συνοχή σημειώνει καθυστερήσεις. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο της έκθεσης, ε, ε, το οποίο θα εμπλωτίσουμε με τροπολογίες, αφορά την εδαφική διάσταση. Η έκθεση επισημαίνει ότι δεν έχουμε πια ε, πολύ ανεπτυγμένες περιοχές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Έχουμε προβλήματα ακόμη και εντός των περιφερειών ε, μεσαίου εισοδήματος. Αλλά ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες υπάρχουν κάποιοι θύλακες, κάποιες ε, ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η, τα προάστια των πόλεων, η περιφέρεια των πόλεων ή ε, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ή οι ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν τα ιδιαίτερα προβλήματα. Και μάλιστα ε, ο Γερμανός πρόεδρος επισήμανε το πρόβλημα της απερίμωσης της υπαίθρου σε πολλές περιφέρειες που από άποψη πλούτου θεωρούνται ανεπτυγμένες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ενώ υπάρχουν και άλλες περιφέρειες που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Το θέμα είναι όμως και σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση του ολοκληρωμένου εδαφικού στόχου. Αλλά πώς ε, θα λάβουμε υπόψη στην πολιτική συνοχής αυτή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων ε, το, και τις ιδιαιτερότητες των, εξόχων, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των ορεινών περιοχών. Γιατί συμφωνώ με την ιδέα να έχουμε λίγους ξεκάθαρους και κοινού στόχους, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να είναι δεόντως ε, διαφοροποιημένη η πολιτική συνοχής, ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε κάποια θεματολόγια που έχουν κάποιους κοινού στόχους, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και κάποιες ενδείξεις στις περιφέρειες ε, για το πώς αντιμετωπίζουν τα ιδιαίτερα τους προβλήματα. Οι εξόχως απόκεντρες, οι δαστικά κέντρα, οι ορεινές περιοχές και ούτω καθεξής. Δεύτερον, οι περιφέρειες που είναι εγκλωβισμένες στην παγίδα του μέσου εισοδήματος του μεσαίου εισοδήματο. Σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοπιστωτική κρίση αποδυνάμωσε τι περιφέρειες από πολλέ απόψει. Σε μερικές περιοχές ε, έχουμε κάποια εδάφη, όχι κατά ανάγκη περιφέρειες, ε, κάποια εδάφη, κάποιες περιοχές που είναι πολύ πιο προηγμένε και κατάφεραν με την καινοτομία να αντιμετωπίσουν την κρίση και επέδειξαν μεγάλη ικανότητα και ανθεκτικότητα, ενώ άλλες ε, περιοχές βρίσκονται σε κάποια πιο δυσχερή φάση ανάπτυξη. Και έχουμε και μία ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών που έχουν πολλές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οπότε είναι δύσκολο να φανταστούμε ανάγκη συνοχής στις περιοχές μεσαίου εισοδήματος. Το θέμα όμως είναι η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών. Και εκεί έγκυται και η παρέμβασή μας με πιο περιφερειακή διάσταση των πολιτικών μας, των περιφερειών. Και εκεί έγκυται και η παρέμβασή μας, ε, με πιο περιφερειακή διάσταση των πολιτικών μας. Και εδώ θα καταθέσουμε επίσης τροπολογίες. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει χωρίς ταμπού να προσεγγίσουμε την ε, επιμέρους περιφέρειες, σε λιγότερο ανεπτυγμένες ή με ειδικά προβλήματα, αν έχουμε μεγάλες αποστάσεις και χάσματα μεταξύ των ε, λιγότερο αναπτυγμένων και των πλέον εύπορων περιοχών, δεν είναι σωστό. Ναι, να έχουμε τις διαφορές, αλλά να μην είναι μεγάλες οι διαφορές και έχοντας επίγνωση της περιπλοκότητας και της ιδιαίτερης του ιδιαίτερα πολυσύνθετου προβλήματος που έχει αυτός ο κατακαιρματισμός και αυτές οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Και σίγουρα οι περιφέρειες μεσαίου εισοδήματος είναι αυτές που χρήζουν μεγαλύτερη στήριξη για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Φορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Φυσικά είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής είναι αλληλένδετα και αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους, πρόκειται φίλονται σε κάποιες βιομηχανικές αλλαγές και θα πρέπει να προσελκύουμε και τις και επενδύσεις σχετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Το λέει στις αιτιολογικές σκέψεις ο εισηγητής. Καλό θα ήταν αυτή την σκέψη να τη μεταφέρουμε και στο διατό. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να, και θεμητό να χρησιμοποιήσουμε κάποιους συμπληρωματικούς δείκτες και είναι σημαντικό αυτοί οι συμπληρωματικοί δείκτες να είναι εύρωστοι, να στηρίζονται δηλαδή σε ενοποιημένα στοιχεία, να λαμβάνουν υπόψη και τις τάσεις, ε, όπως ε, το ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό ανεργίας νέων ή και άλλα κοινωνικά κριτήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για των νέων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως ε, συμπληρωματικοί δείκτες. Το θέμα τώρα της συμπληρωματικότητας μεταξύ της πολιτικής συνοχής συμπληρωματικότητα, γιατί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων χρηματοδοτεί κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και κάποιες δημόσιες επενδύσεις, αλλά ε, να, να αποφέρουν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και που ε, και στον πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα των σχεδίων. Και τέλος, το θέμα της απλούστευσης. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτό ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, το σύμφωνο για τη μεθοδολογία, να έχουμε κάποια βασικά και ουσιώδη στοιχεία που θα πρέπει να που μερικές φορές γίνονται. Πάντως, σίγουρα ε, το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την υποβληθή πριν την, ε, τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα πολιτική συνοχή. Αυτά και σίγουρα στενό χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής αναφέρει επιγραμματικά κάποια θέματα χωρίς να τα αναπτύσσει όμως την έκθεση του. Αυτό οφείλεται στο όριο λέξεων ε, τροπολογιών ε, να καταφέρουμε να αναπτύξουμε αυτά τα θέματα που αναφέρονται ήδη. Γι' αυτό και είπα, λέει η κυρία Μπρέσο, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις τροπολογίες του ε, εισηγητού. Ο κύριος Τόμας έτσι έχει το λόγο. Η κυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τις, ε, την καινοτομία, την ενέργεια, τη μετανάστευση, την ανάπτυξη των πόλων και ούτω καθεξής. Είναι αναφυσβήτητο ότι η οικονομική και χρηματοπιστική κλίση διέκοψε δεκαετία σταθερής ανάπτυξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσε τις ανισότητες μεταξύ των ε, τις χώρες πριν την, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την ε, χρηματοπιστωτική κρίση είχαμε σχετικά ε, χαμηλότερο εισόδημα ε, κοντά στο μεσαίο προϋπολογισμό. Βέβαια, ε, στο μεταξύ αναπτυγμένες περιφέρειες αναπτύχθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς, ενώ συμφωνώ με τις προτάσεις του εισηγητού, γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η πολιτική συνοχής μετά το 2020 να ε, γίνει το πιο αξιόπιστο χρηματοδοτικό μέσο για, για όλες τις περιφέρειες, ώστε να μην ε, ε, μείνουν ανήμπορες μπροστά στην κρίση ή στην παγκοσμιοποίηση ή στις αλλαγές τις τεχνολογικές. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη επενδύσεων σε σχολεία που και ενδιαφέρονται και είναι σε θέση να απορροφήσουν κονδύλιο. Πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό το στοιχείο που αναφέρατε στην παράγραφο 14, την φορολογική και κοινωνική σύγκληση στην εσωτερική αγορά. Είστε Γάλλος. Ε, νομίζω ότι αποτυπώνει το πνεύμα του Μακρόν. Η... Να παραμείνει τουλάχιστον ως έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους συντονιστέ λέει πρόεδρος, και θα συνεχίσουμε με τα μέλη. Παρακαλώ. Στην Ολομέλεια, πριν την παρουσίαση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να έχουμε προχωρήσει κι εμείς, να πάμε πολύ... Έχει κάνει με τη συζήτηση των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων αν το σκεφτείτε περισσότερο, και στα θεματικά. Στην Ολλανδία, γιατί αναφερθήκατε, που είναι καθαρός εισφορέας, ε, συσφορες φορές μέλη. Για διάφορα προγράμματα, για άσπερ και άλλα. Ακόμα και για τις... δηλαδή. σε αυτή την περίοδο και το λέει. Και με τα 7 χρόνια που έχουμε, πολλές φορές στο τέλος έχουμε ξεχάσει που βρισκόμασταν στην αρχή. Θα ήταν λοιπόν πολύ προτιμότερο να έχουμε αυτή την ευελιξία. και να πούμε ότι ξεκινάμε με μία νέα περίοδο. Να δούμε τα κριτήρια, τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει η έκθεση, ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό μείγμα. Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση του ΕΠ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. και μετά ενδεχομένω να προχωρήσουμε σε διαφοροποίηση. Θέλω να πω, πάση περιπτώσει, ότι κάπως απογοητεύτηκα από την έκθεση και την ΕΜΕΝ λέει για την συνοχή, πώς εφαρμόζεται κτλ. Αλλά όσον αφορά το μέλλον, θα ήθελα να είχα δει περισσότερα για το προς τα πού πρέπει να πάμε περισσότερα για συνέργειες με το Horizon για παράδειγμα ή το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε και άλλα πράγματα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και γι' αυτό ξεκίνησα με την ευελιξία που έλεγα ότι κάποιες χώρες τις τη χρειάζονται στον τομέα της γνώσης. Για παράδειγμα. Αλλά και και σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών για την ψηφιακή οικονομία. Και έτσι θα μπορούσε να πετύχει. Αλλά πρώτα πρέπει να ξέρουμε με τι συνδέεται η συνοχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Αν έχεις μια ολοκληρωμένη πολιτική, όπως λέμε ότι είναι η συνοχή τώρα, πρέπει να έχεις και καλά αποτελέσματα. Έτσι κι πάντα χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Ναι, υπάρχει συνοχή στη συνθήκη, δεν μπορεί να μειωθεί η χρηματοδότηση. Όντως χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και έτσι ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για την επόμενη περίοδο. Συμπεριλαμβάνοντας αυτή την ιδέα της ευελιξίας, όπως σας είπα και πριν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μαλέτιτς, ε, κεφάλαιο. Σε αυτές τις περιφέρειες που έχουν παγιδευτεί σε ενεργειακή ένωση και τα άλλα μεγάλα σχέδια, αλλά αυτό που αναφέρετε κι εσείς στην έκθεσή σας, στην κοινωνική διάσταση, οικονομία, για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας δεν θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε ε, τη φτώχεια ούτε να την μειώσουμε. Αντί να μειωθούν, παρά το στόχο που έχουμε θέσει, είχαμε μια αύξηση κατά 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που εξειδίκευσης και χαίρομαι πολύ που το συμπεριλαμβάνετε στην έκθεσή σας, το θέμα αυτό. Πρέπει όμως να τονιστεί αφικών επενδύσεων. Ποια θα είναι η μορφή δηλαδή αυτής της εξειδίκευσης. Θα είναι τμήμα της ε, κάθε θεματικής προτεραιότητας ή θα αποτελεί και είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί, να το συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό. Θέμα που, που είναι πολύ και αυτό ένα στόχο και μια κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Καθώς συζητούμε την 7η έκθεση Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν ήδη προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και το σημαντικότερο πρόβλημα βεβαίω είναι η έγκριση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Λόγω της καθεστέρησης έχουμε μπει στα χαρτογράφητα άδυτα, όχι μόνο γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η μορφή αυτού του πι αλλά διότι δεν ξέρουμε αν και ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα θέσει το επόμενο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια θα είναι η σύνθεση και οι στόχοι της επόμενης Κομισιόν ε, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στους στόχους που σήμερα συζητούμε. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν τρεις αναλλακτικές που έχουν προταθεί για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής είναι σημαντικό και τα τρία σενάρια να αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων της πολιτικής συνοχής στα κράτη-μέλη και την πολιτική υποστήριξη της πολιτικής συνοχής. Γνωρίζοντας ότι στους καθαρούς συνεισφέροντες η πολιτική υποστήριξη περίπτωση στην Ανατολική Γερμανία να μην παραληφθούν ε, κονδύλια συνοχής μετά το 2020. Αυτό οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά είναι σοφό, είναι εύλογο πρώτον για τη Γερμανία και σε δεύτερη λαϊκιστικά, αλλά εκφράζουν αντίθετες απόψεις με, τις, με τα βασικά τους ε, οικονομικά συμφέροντα. Ακούμε απόψει γιατί να δίνουμε ε, πρόσθετα χρήματα ε, στις ανατολικές χώρες, δεν θα πληρώσουμε τίποτα άλλο. Και τα με την έκθεση Μπινκόφσκα, όπου αναφερόταν και αναγνωρίστηκε επίσημα από την Κομισιόν η έκθεση αυτή, ότι από τους καθαρούς συνεισφέροντες κάθε ευρώ που πηγαίνει στην Ανατολή 67% πηγαίνει στη Γερμανία. Και η κατάσταση είναι σταθερή και δεν έχει αλλάξει έκτοτε. Το αντίθετο, οι πρόσφατες εκθέσεις επιβεβαιώνουν την τάση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι από τις χώρες που είναι έροντες, αν και εσείς μέσω συμβουλευτικής και άλλων υπηρεσιών καταφέρετε να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς. Προφανώς η πολιτική συνοχής έχει, είναι αμοιβαία αποφελής και για τις χώρες που συνεισφέρουν και για τις χώρες όψεις που ακούστηκαν ότι θα δίνουμε λεφτά μόνο στις πολύ φτωχές περιφέρειες. Είναι ανοησία ακόμα και για τις πλούσιες περιφέρειες μια τέτοια. Στο όμως τα πράγματα περιπλάκησαν περισσότερο. Ακριβώς γιατί τα κράτη-μέλη έδειξαν μια μεγάλη προθυμία να, που, θα, που, που μας απομένουν το 2021, δηλαδή έως το 2021 όταν και θα εγκριθεί το νέο ΠΔΠ, δεν έχουμε όλο αυτό το διάστημα για απορρόφηση κονδυλίων. Και τέλος, διοικητική ικανότητα. Έχω και της πολιτικής συνοχής. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη στα κράτη-μέλη ώστε... η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξει την πολιτική συνοχής για να μπορέσει ε, να φέρει τα επιθυμητά και αναμενόμενα αποτελέσματα.